Ήλων, ε, Ανά πάσα στιγμή. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε λάβει κάποια μέτρα για να είμαστε σε θέση να συζητήσουμε το 2013. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, θέλετε να προσθέσετε κάτι. Έχετε δικαίωμα να κλείσετε εσείς τη συζήτηση. Όχι. Ωραία λοιπόν. Πολύ καλά. Εξαντλήσαμε και το θέμα αυτό. Λύεται η συνεδρίαση. Συνεχίζεται αύριο το πρωί από τις 9 έως τις 1 συνεδρίαση και από τις 3 έως τις 5 το απόγευμα. Η ημερήσια διάταξη έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Λύεται η συνεδρίαση και καλή ξεκούραση σε όλους.